Θα ξεκινήσουμε στις 8.30 τη συνεδρίαση. Μετά ε, θα υπάρχει ε, μια μέχρι τις 2.30 ε, και μετά θα ξεκινήσουμε πάλι στις 3 μέχρι τις 11. Τελειώνει η σημερινή συνεδρίαση. Σας εύχομαι καλή νύχτα.